Buenos días. Καλημέρα σας. Si les parece, vamos a comenzar. Θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Quería decirles en primer lugar Πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τη συγγνώμη του Προέδρου που κολλείεται σήμερα το πρωί και μου ζήτησε να προεδρεύσω εγώ στην πρωινή μας συνεδρίαση. Πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Για την Αντωνέλα Ροσέτη, συνάδελφο και βοηθό του Πάολο, είναι η βοηθός του συντονιστή της ομάδας μου, του Παύλο Δικάστρο. Είναι η τελευταία της μέρα στην Επιτροπή και όπως ξέρετε η Αντωνέλα πέρασε 11 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επτά από αυτά ως βοηθός του κυρίου Δεκάστρο και ασχολήθηκε με τα θέματα της γεωργίας ε, και ιδιαίτερα με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Μπροστά τη ε, ανοίγονται νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις και νομίζω ότι εκπροσωπώ το σύνολο ε, της Επιτροπής γιατί έχω την τύχη να είμαι σήμερα ο εκπρόσωπος αυτής της Επιτροπής, να την ευχαριστήσω για, για τον ενθουσιασμό της, την επιμέλειά της, την πολύ μεγάλη εργατικότητά της, να την ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή της στο έργο της Επιτροπής και να της ευχηθώ καλή επιτυχία στο μέλλον. Και στον Πάολο, τι να πω. Συλληπιτήρια, συμπάσχουμε με την απώλεια. Ο κύριος Άγνιου. Επειδή και εγώ μπορεί να χάσω τη δουλειά μου, να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως βοηθός. Bueno, está bien. Γιατί όχι. Εντάξει, αποχαιρετούμε βέβαια την Αντωνέλα, αλλά το κάνουμε μη τι άλλο με χιούμορ θα έχουμε νέες φάσεις ζωή για πολλούς. Περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης τώρα, την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, που διακρίνεται σε διάφορα στάδια. Είχαμε μετά την ψηφοφορία της εντολής για τον τριμερή διάλογο, την εκπόνηση της γνωμοδότησής μας για το γενικό προϋπολογισμό. Επίσης, επεξεργαζόμαστε κάποιες τροπολογίες για τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία του προϋπολογισμού. Μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2017 και μας ε, το μεταβίβασε μόνο την 1η Ιουλίου. Και οι εκτιμήσεις του Συμβουλίου θα μοιραστούν στα μέσα Ιουλίου, όχι νωρίτερα. Πολλέ Τροπολογίε Επιτροπή Γεωργίας ε, για τι διάφορε δημοσιονομικέ γραμμέ ε, σχετίζονται με τι εκτιμήσει ε, και τι προβλέψει του Συμβουλίου. Οπότε σήμερα ο εισηγητή μα ο κύριο Γιάρ δεν θα μα δώσει αριθμητικά στοιχεία από την γνωμοδότηση, αλλά θα μα κάνει μια γενική παρουσίαση. Επίση ο κύριο Γιάρ κατέθεσε μια έκθεση για το Γενικό προπολογισμό του 2017 με βάση το προσχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την γνωμοδότηση αυτή θα μας την παρουσιάσει αμέσως ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε στην πολύ καλή σας εισαγωγή, λόγω του Brexit ο χρόνος αρχίζει να πιέζει, διότι τα νούμερα της Κομισιόν ήρθαν πολύ καθυστερημένα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα πρώτα απ' όλα, διότι τα συμπεράσματα θα είναι δύσκολα, 30 Αυγούστου η Επιτροπή Προϋπολογισμών όχι, περιμένετε. Ναι. Ναι, έχετε δίκιο. 30 Αυγούστου ε, είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών και μετά το Σεπτέμβριο θα ψηφίσει το έγγραφο. Το Σεπτέμβριο και μετά η υιοθέτηση θα γίνει στην ολομέλεια, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε ήδη από τις 29 Αυγούστου να κάνουμε μια συνεδρίαση μεταξύ συγκητών και σκιωδών. 29, <clears throat> συγγνώμη, 29 Αυγούστου βέβαια δεν έχουμε άλλη δυνατότητα για να συναντηθούν σκιώδης και εισηγητής για να συζητήσουμε τα πράγματα της ουσίας. Αυτά τα ε, έχω γράψει και σε email. Δεύτερη προκατακτική παρατήρηση. Με εκπλήσουν κάπως οι σκιώδεις εισηγητές που έχουν ήδη εγκύψει στο σχέδιο και διαπιστώνουν ότι λείπουν τρεις παράγραφοι. Δεν τις διαγράψαμε διότι μας φάνηκαν ασήμαντες, αλλά απλώς το κείμενο ήταν υπερβολικά μακροσκελές. Γι' αυτό βγάλαμε τρεις παραγράφους. Μπορούμε όμως να τις επαναφέρουμε, διότι αυτό επιτρέπεται, μέσω τροπολογιών. υποκληθήκαμε, αν θέλετε, λίγο στους κανόνες που επιβάλλει η διοίκηση. Περικόψαμε λίγο το κείμενο στην πρώτη εκδοχή του, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Και γι' αυτό επιθυμώ να καθησυχάσω τους σκιώδεις συζητητές. Για την ίδια τη γνωμοδότηση τώρα. Στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύγκριση με το 2016, οι κατανομές μειώνονται κατά 7,6%. Οι περικοπές στον πρώτο πυλώνα τις λαμβάνουμε υπόψη διότι αναμένονταν άλλωστε στον πρώτο πυλώνα πέφτουμε αρκετά μέσα στο στόχο γνωρίζουμε και πόσο υψηλές είναι οι πληρωμές οι περικοπές αυτές προβλέπονταν έχουν σχέση και με δημοσιονομική τεχνική διότι μπήκε και η Κροατία δεν είναι όμως εκεί τα μεγάλα προβλήματα νομίζω ότι μπορούμε απλώς να λάβουμε γνώση διότι οι άμεσες ενισχύσεις είναι εξασφαλισμένες και στο ύψος που απαιτείται. Για τις άμεσες ενισχύσεις δεν, δεν χρειαζόμαστε αποθεματικό, διότι είναι ξεκάθαρα τα νούμερα και είναι σίγουρα. Στην παράγραφο 3 έχουμε 23% μείωση, κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε ως έχει, ή εν πάση περιπτώσει έχουμε ανάγκη από κάποια αιτιολόγηση και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και από την Κομισιόν. Δύο προσπάθειες εξηγήσεως δίνονται εδώ. Όπως είπα, αφενός οι περικοπές την από, μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Δεύτερο, όταν εξετάσει κανείς την τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, υπάρχει καμπύλη που διαγράφω και με το χέρι, και που θα σημαίνει ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα χρειαστεί να δεχτούμε περικοπές. Όμως όπως είναι τώρα δεν μπορούμε να τη δεχτούμε διότι ο δεύτερος πυλώνας είναι σημαντικός για την ανάπτυξη πέθρου και ιδίω για ε, επενδυτικά προγράμματα. Τρίτο, ε, μας, μας ενοχλεί η περικοπή κατά το ίμιση του περιθωρίου, διότι έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι έχουμε ήδη χαμηλότερο περιθώριο σε σχέση με τα προηγούμενα σχέδια προϋπολογισμών και γιατί de facto το περιθώριο είναι και ένα μικρό αποθεματικό για απρόβλεπτα, ιδίω για κρίσεις. Γι' αυτό λέμε ότι πρώτον θέλουμε να παραμείνει το περιθώριο, δεύτερον να μην περικοπεί, τρίτον είμαστε απολύτως αντίθετοι το περιθώριο να διατεθεί σε άλλους τομείς. Και θα διεξαχθούν και έντονε συζητήσεις και στην Επιτροπή Προπολογισμών. διότι ζητούν να μειωθεί το περιθώριο και να δοθούν ορισμένα από τα χρήματα αυτά για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Οι χώρες μέλη, ωστόσο, οφείλουν να κατεβάσουν άλλε ιδέες για την αντιμετώπιση του κόστου του προσφυγικού. Δική του υπόθεση είναι δεν μπορούμε να δεχθούμε εμείς να βάλουν χέρι στον προπολογισμό της ε, γεωργίας. Υπάρχουν και καλά πράγματα. Περισσότερα ε, χρήματα για, τη, για τους συνεταιρισμούς παραγωγών, για τη μελισσοκομεία επίσης. Ναι, η βασίλισσα των Μελισσών έχει αποχωρήσει από το κοινοβούλιο, αλλά για τη μελισσοκομεία δίνονται περισσότερα χρήματα. Αυτό μα ικανοποιεί. Πρέπει να βρεθεί για καλύτερο monitoring για την κρίση, για να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Πρέπει, όπως είπα, να διατηρηθεί το περιθώριο. Και στην παράγραφο 14, για να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Γεωργία, και το ΦΕΟΓΑ. Χρειάζεται λοιπόν ο προπολογισμό του ΦΕΟΓΑ. Όμως, όταν αυξάνονται οι απαιτήσει απέναντι στη γεωργία, η κοινωνία δηλαδή έχει όλο και περισσότερες προσδοκίες από τη γεωργία, οφείλει εδώ η γεωργία να ανταποκριθεί, αλλά παρακαλώ πολύ να τις προσφερθούν και τα δημοσιονομικά μέσα. Όποιος έχει παραπάνω επιθυμίες και προσδοκίες πρέπει να βάλει και το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Αυτά είναι λίγο πολύ τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Το μεγάλο σημείο διαφωνίας είναι οι περικοπές, ιδίω στον δεύτερο πυλώνα, που δεν είναι και τόσο εύκολο να αποδεχτούμε. Αναμένω βεβαίω με ενδιαφέρον την περαιτέρω συζήτηση. Χαίρομαι ήδη για τη συνεργασία με του κοιόδη και αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε τον ίδιο τρόπο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε. Ελπίζω μάλιστα ορισμένα από τα θέματα, ορισμένα από τα σημεία μας να μπουν και στην έκθεση της Επιτροπής των Υπολογισμών. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρου του Τίμπορ παρεμβαίνω του συναδέλφου που είναι σκιώδη συζητητή και ο οποίο σήμερα δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ μαζί μα. Απλά για να πω ότι ευχαριστώ τον Πέτερ για τι προσπάθειέ του. Ε, είναι απόλυτα συντονισμένα σε εργασίε του. Οι ανησυχίε είναι πολλέ. Ε, Όπω είπε ο συνάδελφο Γιάρο, ο κίνδυνο ε, να είναι μεγάλε οι περικοπέ στον προπολογισμό τη Γεωργία ε, επιβάλλει την προσοχή μας, ε, την ιδιαίτερη προσοχή μας για αυτή τη γνωμοδότηση. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε για τις συνεδρίες της 29 η Αυγούστου και τη στρατηγική για τις τροπολογίες, ούτως ώστε να μην περάσει αυτό το υποθετικό σενάριο που μπορεί να προτείνει η Κομισιόν, γιατί θα είναι σημαντικές οι περικοπές. Και ακόμα και η μετατόπιση των πόρων στον προϋπολογισμό για να καλύψουμε άλλα προβλήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά η Γεωργία περνά δύσκολες εποχές. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε να μειωθεί ο προϋπολογισμός της. Ευχαριστούμε λοιπόν Πέτερ και θα συντονιστούμε. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Δεκάστρο. Άλλος κανείς για τον προϋπολογισμό ich möchte mich natürlich auch im Namen unserem Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερο τον Πέτερ Ιά, για τι εξηγήσει που έδωσε. Τον υποστηρίζουμε. Εν πάση δε περιπτώσει πρέπει από κοινού να αναπτύξουμε μια στέρεα στρατηγική, ώστε να μην χρειαστεί να αναμένουμε σημαντικές περικοπές στην Επιτροπή Γεωργίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πραγματικά χρήσιμη γνωμοδότηση με συμμετοχή όλων των πολιτικών ομάδων και εμείς πολύ ευχαρίστως θα συμβάλλουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μίλλερ. Ο κύριος Βιέγας. Καλημέρα σας. Ο προϋπολογισμός αυτός πιστεύω ότι έχει πάρει στραβό δρόμο. Το δρόμο του αργού θανάτου της Γεωργίας. Γιατί έχουμε αφενός μία αλληλουχία μεταρρυθμίσεων της κοινής ε, αγροτικής πολιτικής ε, προς την κατεύθυνση της ε, απελευθέρωσης, αλλά δεν έχουμε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε την αποσταθεροποίηση των αγορών. Και αυτό ανακλάται και στον προϋπολογισμό του 2017, ο οποίος εμπεριέχει αυτή την εσωτερική αντίφαση. Δεν ανταποκρίνεται σε μία αντίξωη πραγματικότητα που δεν την επιθυμούμε, αλλά που είναι φυσική απόρρια των πολιτικών των τελευταίων χρόνων. Ε, είχαμε κατάργηση των ε, γαλακτοκομικών ποσοστώσεων ε, και πρόγραμμα απελευθέρωσης με δραματικές συνέπειες ό,τι αφορά τις απότομες διακοιμάσεις και την αστάθεια των τιμών. Και πέρυσι είχαμε και την εξάντληση όλων των περιθωρίων και όλων των μέσων που στόχο είχαν την αντιμετώπιση αυτής της αστάθειας. Αυτό που διεκδικούμε είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή των κονδυλίων, ώστε να προσφέρουμε κάποια αντιστάθμιση για αυτή την οξύτατη κρίση που βιώνει ο γεωρικός κλάδος αυτή τη στιγμή. Όπως λέγαμε και στο παρελθόν, πιστεύουμε και σήμερα ότι δεν θα πρέπει ο γεωργικός προϋπολογισμός να υποστεί τις συνέπειες του ρωσικού αποκλεισμού, γιατί το ρωσικό εμπάργο ήταν πολιτική απόφαση. Θα πρέπει το σύνολο λοιπόν του προπολογισμού να αναλάβει αυτές τις συνέπειες του πολιτικού μέτρου και να μην πληρώσουν τα σπασμένα οι γεωργοί και ο γεωργικό προπολογισμό. Δεν φταίνει αυτοί για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέβαλε το ρωσικό εμπάργο τα αποτελέσματα του οποίου τα βιώνουμε ακόμη και σήμερα. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα είναι η υγιεινή και των φυτών και η υγεία των ζώων. Γιατί έχουμε όλο και περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς και παράσιτα που ε, επηρεάζουν είτε τα φυτά είτε τα ζώα, ε, τα βοηδή, τα χοιρινά. Πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο αρρώστιες ε, φυτών και ζωονόση που επίσης επηρεάζει την κατάσταση στην αγορά. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κονδύλια για την καταπολέμηση και ακόμη καλύτερα την πρόληψη των ασθενειών στη χλωρίδα και στην πανίδα και τις ε, επιδημιολογικές συνέπειές τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βιέγας. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ μιλάμε για μείωση του προϋπολογισμού της Γεωργίας. Αυτό που μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι ότι πριν δύο μήνες βρίσκομαι σε μια συζήτηση ε, περί δημοψηφίσματος με τον Επίτροπο Χόγκαν. Είναι άλλο ένα θέμα. Πρέπει να συζητηθεί το κατά πόσο έπρεπε να έχει έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να έχει παροτρύνει τον κόσμο στο πώς να ψηφίσει. Το έκανε όντως και εγώ ήμουν κατά αυτού σε μια συζήτηση. Και πήρα ένα ρίσκο και είπα ότι κατά την άποψή μου ο προπολογισμό της γεωργία επρόκειτο να περικοπεί ώστε να βρεθούν κονδυλία για τη μεταναστευτική κρίση και ότι εγώ ανέμενα να απορρίψει όσα είπα ο Επίτροπος αλλά δεν τα απέρριψε το οποίο με έκανε να σκεφτώ ότι μάλλον επρόκειτο να γίνουν τέτοιε περικοπέ. Εγώ κοιτώντα λίγο στο μέλλον, και αυτό δεν έχει να κάνει με τον Brexit, Είμαι εδώ 7 χρόνια και ακούμε διαρκή γκρίνια από αγρότες που θέλουν λεφτά για το ένα και για το άλλο και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επινοήσει κάποιο σύστημα συνταξιοδότησης με αξιοπρέπεια ώστε οι αγρότες οι οποίοι ζουν σε μη βιώσιμα αγροκτήματα να πάρουν κάποιο ανταμοιβή, κάποια αποζημίωση και ε, οι, ε, τα, τα αγροκτήματά τους δεν μπορούν πλέον να, να λάβουν επιχορηγήσεις ε, και να μετατραπούν σε άγριες ή ίσως να τη μεταβιβάσουμε σε ένα νέο γεωργό χωρίς επιχορηγήσεις ο οποίος θα αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές του ικανότητες ή θα καλλιεργήσει λαχανικά για την τοπική αγορά. Κοιτάξτε πόσο είναι το διοικητικό κόστος αυτής της επιχορήγησης των αγροκτημάτων 5 και 10 εκταρίων δεν έχει νόημα. Εγώ ακούστηκα σαν αρετικό λέγοντα κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά το πιστεύω. Ακράδαντα. Σα ευχαριστούμε κύριε Άγνιο. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Να πω κάτι στον κύριο Άγνιο. Εσείς συμμετέχετε πολύ σε αυτή την Επιτροπή και δεδομένου ότι είστε ευρωσκεπτικιστής ε, ε, θα μπορούσαν μερικοί αγρότες να έρθουν εδώ και να παλέψουν για αυτό το έργο. Μου φαίνεται περίεργο που μόνο ευρωσκεπτικιστές έρχονται εδώ. Θα έπρεπε να έρθουν και μερικοί φίλοι της Ευρώπης εδώ για να μαχηθούν για όλο αυτό, όχι αγρότες. Ξέρετε, όλοι έχουμε να κάνουμε μια δουλειά όλη μου τη ζωή προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους ότι είναι καλή ιδέα να λαμβάνουν περισσότερα χρήματα οι αγρότες και αυτά τα χρήματα δεν μένουν στις τσέπες τους, είναι χρήματα που δαπανώνται. Το έχω ξαναπεί σε αυτή την Επιτροπή. Ε, εγώ δεν έρχομαι από αγροτικό παρελθόν. Ο πατέρας μου ήταν ξυλουργός και χωρίς τα χρήματα της ΚΑΠ που ήρθαν σε όλες τις ε, ε, περιοχές μας ε, δεν ε, θα μπορούσαν να είχαν σπίτια ε, και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα. Αλλά το δεύτερο, και ξέρετε θα κοβόταν εντελώς ο προπολισμός αν ακούγαμε ορισμένους, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί κόσμος ενοχλείται που πολλά από αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν καν στους αγρότες τελικά. Πηγαίνουν στους ε, ε, βιομηχάνο μαζική παραγωγή, τον Λάρι Γκούντμαν στην Ιρλανδία, ο οποίο έχει το δικό του ιδιωτικό αεροσκάφο. Πώ δικαιολογεί κανεί έναν προπολογισμό που καταλήγει στι τσέπε ενό ατόμου που έχει δικό του ιδιωτικό τζετ. Δεν μπορούμε να το πουλήσουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε όμω να λειτουργήσουν τα πράγματα και να πάψει να υπάρχει πίεση προ τα κάτω στον προπολογισμό. Πρέπει να του πείσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Ευχαριστούμε κύριε Φλάναγκαν. Ο κύριος Άλμπερτ Ντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 52 χρόνια είμαι. Κάθε χρόνο υφίσταται η Γεωργία επιθέσεις. Όλοι λοιπόν πρέπει να ορθώσουμε μαζί το ανάστημά μας και να προβάλλουμε τα ορθά επιχειρήματα. Έχετε δίκιο ότι τα χρήματα δεν διατίθεται πάντοτε με τον πιο λογικό τρόπο και τον πιο σκόπιμο. Αλλά δεν είναι δυνατόν η γεωργία να χρησιμοποιείται ως υλοτομείο για να τροφοδοτούνται άλλες πολιτικές. Πότε είναι το εμπάργο της Ρωσίας, πότε το ένα, πότε το άλλο, το οποίο επιβαρύνουν εν τέλει την αγροτική οικονομία. Ούτε μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από τον προπολογισμό της Γεωργίας το πρόβλημα των προσφύγων. Σωστά τα είπατε αυτά εσείς οι προηγούμενοι και ευχαριστώ και τον Πέτερ Γιάρ που έχει αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο. Είχα εκνευριστεί κιόλα που πριν από λίγε εβδομάδε είχε ζητήσει ο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών είχε πει μάλλον ότι το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προπολισμού το απορροφάει η Γεωργία. Εγώ είχα πει τότε ότι εάν όλες οι δημόσιες δαπάνες γίνονται αντικείμενο διαχείρισης όπως ο προπολογισμό της Γεωργίας, η διαχείριση αυτή θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερη. Πρόκειται για την ομάδα εκείνη ανθρώπων, ενώ του αγρότες, οι οποίοι τροφοδοτούν με τρόφιμα 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χρήματα που λαμβάνουν είναι άπειρο ελάχιστα σε σύγκριση με το έργο που επιτελούν. Ο προπολογισμό τη Γεωργίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο έφτανε το 87%. Σχεδόν τίποτε άλλο δεν χρηματοδοτούνταν από τις Βρυξέλλες τότε. Μειώθηκε το ποσοστό αυτό, το 1% παραπάνω που μας δώσαν, ε, δεν θα δεχτούμε να μας το πάρουμε πίσω. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντές. Και τέλος ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπέλντερ είναι ο σχεδόν από την ομάδα μου, αλλά κολλείται σήμερα και τον αναπληρώνω εγώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάρ για την ε, αξιολογότατη γνωμοδότησή του. Ε, είναι πολύ ικανός πολιτικός και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Και θα συμβάλλουμε ε, στις περαιτέρω συνομιλίες με τους κοιόδης και τον κύριο Γιάρ. Εγώ θυμάμαι και τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε στου συντονιστέ για τι περικοπέ στη Γενική Διεύθυνση γεωργία. Ίσως ο εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα μπορούσε να το σχολιάσει. Γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, οι αναγγελθήσεις περικοπέ στη Γενική Διεύθυνση γεωργία. Ε, εγώ πρωτεξελέγη το 1999. Τότε η Γεωργία ήταν πάνω από 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού. Τώρα είναι πολύ λιγότερο και συνέχεια μειώνεται. Πιστεύω και εγώ πως και προλαλήσαντες ότι έχουμε καθήκον και ευθύνη σε όλα τα επίπεδα να πιάνουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων και να αξιοποιούνται σωστά. Αλλά είναι σημαντικός ο γεωργικός προπολογισμό. Άσχετα με την έκβαση του Βρετανικού δημοψηφίσματος και για την επόμενη διετία το δύσκολο θα είναι για τον κύριο Άγνιου να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στους γεωργούς ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ καλύτερα. Εμείς πιστεύουμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισχυρότερη η γεωργία και θα είναι καλύτερα. Για να δούμε πώς θα τους πείσετε τώρα και πώς θα τηρήσετε τις υποσχέσεις σας. Κάθε φορά ακούμε την πρόταση για περικοπές το θέμα είναι να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων. Το θέμα είναι τα χρήματα να φτάνουν στους άμεσα ενδιαφερόμενους, είτε για την αγροτική ανάπτυξη, είτε για τις άμεσες ενισχύσεις. Πολύ εύστοχο το σχόλιο του κυρίου Φλάναγκα και το διαπιστώνω και στην εκλογική μου περιφέρεια. Τα γεωρικά κονδύλια στηρίζουν την αγροτική οικονομία. Γιατί αν δεν είχαμε αυτά τα κονδύλια στην αγροτική οικονομία μέσω του γεωρικού προπολογισμού, τι θα κάναμε. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούν σαν καραμέλα την έννοια της επιδότησης, επιχορήγησης, αλλά δεν είναι μια επιχορήγηση που βγαίνει στον Γεωργό για να παράγει, αλλά είναι επιχορήγηση και για τον καταναλωτή. Γιατί αν δεν λάβει αυτά τα χρήματα, αυτέ τι επιδοτήσει ο Γεωργό, πώ θα καλλιεργήσει ε, τα χωράφια του να παράγει τρόφιμα και να γεμίσουν τα ράφια το σούπερ μάρκετ με τρόφιμα για να μπορεί να αγοράζει ο καταναλωτή. Και τα φθηνά τρόφιμα έχουν ένα άλλο χειρότερο τίμημα. Θα το πληρώνουμε διπλά. Αυτό θα κάνουμε από τις υπερβολικές οικονομίες, γιατί η παραγωγή ποιοτικών τροφίμων είναι δαπανηρή. Πρέπει να πληρώνουμε τον Γεωργό Αξιοπρεπός, γιατί αν παράγει σε τιμές κάτω του κόστους, πρέπει αμή τι άλλο να λαμβάνει κάποια αντιστάθμιση, κάποια αποζημίωση, κάποια επιδότηση. Και Ίσως έτσι είχε καλύτερη κατανόηση ο καταναλωτής και να, να γνωρίζει ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η παραγωγή τροφίμων. Γι' αυτό και θα πρέπει να μείνετε αξιοπρεπώς ο Γιώργος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νίκολσον. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο, στον κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε. Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να αναπτύξω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα, γνωρίζετε βέβαια το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο που υπαγορεύει ότι υποβάλλεται το σχέδιο προϋπολογισμού με κάποια καθυστέρηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ε, επιφέρει κάποιες συνέπειε, πρακτικές συνέπειε και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο βεβαίω σε ό,τι αφορά τη σύνταξη τη γνωμοδότησής σας για τα επιμέρους θέματα που έθιξε ο εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής σας τώρα. Και πρώτα εισαγωγικά. Η τέχνη στη σύνταξη του προϋπολογισμού είναι ο ακριβής σχεδιασμός των δαπανών του επομένου έτους. Δεν έχει πολύ νόημα δηλαδή για όσους συντάσσουν τον προπολογισμό να εγγράφουν υψηλά ποσά στον προϋπολογισμό του 2017 εάν γνωρίζουμε από τώρα ότι τα, τα ποσά αυτά δεν πρόκειται να δαπανηθούν. Έτσι πρέπει να κανείς να εξετάσει προσεκτικότερα αυτές τις δίθεν περικοπές. Πρώτα για το περιθώριο. Ένα μέρος του περιθωρίου στην κατηγορία 2, που είναι διαθέσιμο στην κατηγορία 2, σχεδιάζεται να διατεθεί για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Αυτό έγινε διότι θεωρούμε, εξ όσων γνωρίζουμε σήμερα, ότι τα ποσά αυτά δεν θα απορροφηθούν στην Γεωργία στο έτος 2017. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι μπορούν και πρέπει να διατεθούν για την αντιμετώπιση αυτών των σημαντικών κρίσεων. Για τα επιμέρους τώρα θέματα που αναφέρατε, ο προκυπευτικά, το γάλα που διατίθεται στα σχολεία. Και εδώ πάλι περιγράφεται περικοπές που έχουμε εγγράψει στον προϋπολισμό, αλλά αυτές εκκινούν πάντοτε από τα όσα γνωρίζουμε σήμερα και από την εκτέλεση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Οι χώρες μέλη, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν είναι καν σε θέση να δαπανίσουν περισσότερα για το 2017 από αυτά που έχουμε ήδη εγγράψει στον προϋπολογισμό. Δεν έχει λοιπόν πολύ νόημα να εγγράφουμε υψηλότερα κονδύλια στον προϋπολογισμό εάν γνωρίζουμε εκ τον προτέρων ότι δεν πρόκειται να απορροφηθούν τα κονδύλια αυτά, διότι εν τέλει θα χαθούν τα χρήματα αυτά για την αγροτική οικονομία εάν δεν έχουν δαπανηθεί όντως μέχρι τον Οκτώβριο του 2017. Μια σύντομη προσπάθεια εξηγήσεως για τον πυλώνα 2 για τη στήλη 2. Είπατε ότι και εκεί θα γίνουν περικοπές. Ωστόσο, το 2016 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος στην ανάπτυξη της υπέθου Υπάρχουν πάντοτε επικαλύψεις ανάμεσα στα δύο δημοσιονομικά πλαίσια και αυτό ισχύει για το 2016, δηλαδή τα προγράμματα 2007 έως 2013 εξακολουθούσαν, τα προγράμματα αυτής της περίοδου δηλαδή, να λειτουργούν και πρόβλεπαν πολλές δαπάνες. Ταυτόχρονα αρχίζουν τα προγράμματα του 2014-2020. Αρχίζουν ήδη λοιπόν να λειτουργούν από το 2016. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αυτό που συνέβη είναι ότι πληρωμές που προβλέπονταν κανονικά το 2014 και ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα κατανείμαμε στα έτη 2015 και 2016 για να προσφέρουμε στις χώρες μέλη την αναγκαία ευκαμψία ή ευελιξία για να συνεχίσουν τις πληρωμές των παλαιών προγραμμάτων. Υπάρχει λοιπόν μια ιδιαίτερη κατάσταση και ιδίως για το 2015 και 2016, ιδίως για το 2016. Και αυτό που προτείνουμε στον προπολογισμό του 2017 είναι στην ουσία μια επιστροφή στην ομαλότητα. Δηλαδή η ομαλή εκτέλεση των προγραμμάτων αρχίζει και προχωρεί που σημαίνει ότι προβλέπονται 14 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Και αυτά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ ούτως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 17. Και θεωρούμε ότι αυτό ανταποκρίνεται σε ομαλές συνθήκες. Όπως είπα, 14 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι αυτά που προβλέπονται για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται πραγματικά για περικοπές, απλώς εισερχόμεθα πλέον πάλι σε, μια, ένα φυσιολογικό καθεστώς και εξαλείφουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα το, του πλαισίου 2007 έως 2013. Άρα, κατά τη γνώμη της Κομισιόν, δεν είναι πραγματικές περικοπές αυτές στον τομέα της ε, γεωργίας. Θεωρούμε ότι ο προπολογισμό που έχουμε καταθέσει είναι ρεαλιστικός. Καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα για το έτος 2017. Γνωρίζετε όμως βεβαίως επίσης ότι δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί το 2017. Το φθινόπωρο, και θα συζητηθεί άλλωστε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχουμε πάλι την ευκαιρία με διορθωτικό προϋπολογισμό να προβλέψουμε δαπάνες για ενδεχόμενες κρίσεις. Και γνωρίζετε ότι την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών θα γίνει συζήτηση και θα υποβληθούν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν είναι απαραίτητα νέα κονδύλια, θα έχουμε τη δυνατότητα με τη διορθωτική επιστολή του Σεπτεμβρίου να προτείνουμε τα συγκεκριμένα κονδύλια στα πλαίσια της κατηγορίας 2. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις, τις εξηγήσεις. Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή της γνωμοδότησης, τον κύριο Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, σκιώδης για τη συνεργασία τους, ευχαριστώ για τη συζήτηση και ευχαριστώ και τις εξηγήσεις από πλευράς Κομισιόν. Βεβαίως πρέπει να προσέξει κανείς, το απευθύνω αυτό στους συναδέλφους μου, μιλούμε για τον προϋπολογισμό του 2017. Έχω και πολλές ιδέες για βελτίωση της αγροτικής μεταρρύθμισης, αλλά μιλούμε εδώ για τον προπολογισμό του 2017, επαναλαμβάνω, που σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιες συνθήκες ισχύουν εκεί. Για την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής ξανακαταστήσαμε σαφείς τις ιδέες μας. Τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα η Γεωργία, έχει εμφανιστεί και ως αξιόπιστος εταίρος στην ε, διαχείριση του προϋπολογισμού και μάλιστα χωρίς καν να τα αντιληφθεί αυτά η κοινή γνώμη έχουμε μειώσει το ύψος του αγροτικού προϋπολογισμού και κατά κεφαλήν. Αυτό είναι σημαντική επιτυχία και το λέω και με αυτοπεποίθηση. Η Γεωργία μας θα ήταν σούπερ ευχαριστημένη αν είχαν επαρκέ εισόδημα από τις τιμές τη αγορά χωρίς να χρειάζονται καμία απολύτως παρέμβαση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, επειδή του επιβάλλονται κανόνε κανόνες, έχουν και αυτή απέτηση για κάποια αντιστάθμιση. Το ποσοστό του αγροτικού προϋπολογισμού στον ευρωπαϊκό συνολικό προϋπολογισμό μειώνεται διαρκώς. Οι γεωργοί αποδείχνονται πραγματικά αξιόπιστε τέρι. Δεν είμαστε διόλου ο πίθος των Δαναίδων που καμιά φορά μας παρουσιάζουν. Για το περιθώριο έχουμε κάνει τη σχετική εκτίμηση. Ένα τμήμα των χρημάτων αυτών θα πάει για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ξέρουμε βεβαίως ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όμως στον τριμερή διάλογο θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη αρχή, δηλαδή αυτός που ζητεί κάτι πρέπει και να πληρώνει, δηλαδή οι χώρες μέλη. Οι δαπάνες για το προσφυγικό βασίζονται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να βάζουν χέρι στον ήδη πολύ αυστηρά ορισμένο δικό μας προπολογισμό. Τα άλλα για τη δεύτερη κατηγορία, αυτά, σημειώνω αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για τεχνικού χαρακτήρα κίνηση, θα τα περιλάβουμε ίσως σε μια ωραία τροπολογία. Και βεβαίως γνωρίζουμε και τι γίνεται στις χώρες μέλη. Όταν τα πρώτα χρόνια δεν απορροφώνται τα χρήματα των προγραμμάτων, στο δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή, καμιά φορά ξεχνούν οι χώρες μέλη ότι πρέπει να διαθέσουν αργότερα περισσότερα χρήματα. θα προσπαθήσουμε σε ένα shadow meeting να περιλάβουμε τις διάφορες ιδέες των συναδέλφων, τα έχω σημειώσει αυτά και χαίρομαι εν αναμονή της περαιτέρω καρποφόρου συνεργασίας. Πιστεύω ότι θα είναι τελικά μια χρήσιμη γνωμοδότηση που ελπίζω να υποστηριχτεί από μεγάλη πλειοψηφία, σημαντικό αυτό, εάν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι μέσω του αγώνα μας υπέρ της αγροτικής οικονομίας, και τελικώς να καταλήξουμε σε μια ε, στέρεη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Σίγουρα εν τη ενός ίσχυς. Και μόνο συσπηρωμένοι θα καταφέρουμε κάτι. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στις 22 Ιουλίου 2016 στις 12 το μεσημέρι. Τότε έλεγε η διορία για την υποβολή τροπολογιών που πρέπει να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά. Για σας πανεύκολο το εγχείρημα κύριε Άγνιο. Εμείς αγαπούμε και τα αγγλικά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο στα αγγλικά λοιπόν μπορείτε να υποβάλλετε τι τροπολογίε σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις 22 Ιουλίου. Επόμενο σημείο τη ημέρησης διάταξη, το σημείο 10 έχει αναβληθεί για τη συνεδρίαση της 26 Σεπτεμβρίου. Μας ενημέρωσε χθε σχετικά ο Πρόεδρος. Οπότε περνάμε κατευθείαν στο σημείο 11 την παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, των εξελίξεων ε, για την ε, αρρώστια των φυτών, το βακτήριο Ξυλέλα φαστιδιώσα. Το πρώτο, κρούσμα, το πρώτο της ξυλέλαφας στη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 στην Νότιο Ιταλία. Το βακτήριο αυτό ε, προσέβαλε αρκετές χιλιάδες εκτάρια ελαιώνων στην περιοχή της Απουλίας. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει μέτρα για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας αυτής που προσβάλλει τα δέντρα και τα νεκρώνει με αργό ρυθμό. Το τοπικό περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο του Λάτσιο υιοθέτησε νομικά μέτρα που ανέστηλαν την εντολή απομάκρυσης των δέντρων και φυτών που βρίσκονταν κοντά σε μολυσμένα ελαιόδεντρα και έθεσε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με θέμα την εγκυρότητα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 9 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, δημοσίευσε την απόφαση του με την οποία επιβεβαίωνε την εγκυρότητα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την οδηγία του Συμβουλίου 2000-29 ε, ερμηνεύοντάς την υπό το φως των αρχών της προφύλαξης και της αναλογικότητας. Στη συνεδρίαση των συντονιστών της 21ης Ιουνίου αποφασίστηκε η οργάνωση μιας ανταλλαγής απόψεων με εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΤΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις αυτού του βακτηρίου και την εξάπλωσή του, της ξυλέλα φαστιδιώσα. Και μάλιστα στείλαμε και πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος για συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αρχικά ήταν ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Μπέρναρ Φανγκέτε. Τελικά, δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Θα μας ενημερώσει η κυρία Ντόροθι Άντρε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και τα μέτρα που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας αυτής στη Νότια Ευρώπη. Μετά την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε ερωτήσεις ή να κάνετε παρατηρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Αντρέη που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα στους κύριε και κυρίες ευρωβουλευτές. Ε, Ζήτω συγγνώμη εκ του Μπερνάρ Μαγκουτέν του διευθυντή μου που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το σημείο στην κόμμα Άγκρη. Να σας παρουσιάσω την τρέχουσα κατάσταση, το τι συνέβη από τότε που ο Επίτροπος Καΐτης ήρθε στην Επιτροπή αυτή κατά τη διάρκεια του διαρθρωτικού διαλόγου στις 15 Μαΐου, όπου εξήγησε ότι η Κομισιόν έπαιρνε φυσικά πολύ στα σοβαρά αυτή την ασθένεια και μεριμνούσε ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μέχρι σήμερα τρία από όλα τα κράτη-μέλη έχουν ανοιχνεύσει την παρουσία της ξυλέλαφας στην επικράτειά τους. Η Ιταλία, το 2013, η Γαλλία το 2015 και πολύ πρόσφατα η Γερμανία. Θα σας αναπτύξω και τις τρεις περιπτώσεις. Ε, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει επιτήρηση της επικράτειας και η επιτήρηση του 2015 έδειξε ότι δεν υπήρχε εξελέλαφες δύο της επικρατείε τους. Από το Μάρτιο λοιπόν και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε για νέες αιστείες στην Ιταλία. Η Κομισιόν επίσης και κάνει και κάποιον έλεγχο. Η Ιταλία γνωστοποίησε στην Κομισιόν ότι ένα κόμμα της επικράτειας θεωρείται ότι είναι απαλλαγμένο από την ξυλέλα και βάσει αυτών των διαφορετικών στοιχείων η Κομισιόν έθεσε σε ψήφο 15 Απριλίου μια απόφαση που αλλάζει την οριοθετημένη ζώνη κατά 40 χιλιόμετρα προς τα πάνω, εξαπλώνοντας κατά 40 χιλιόμετρα προς το βορρά. Κάτι που επιτρέπει ουσιαστικά στην περιοχή του Λέτσε να υπάρξει ε, εξαφάνιση και όχι εκρίζωση της ε, ασθένειας ε, και υπάρχουν δύο ζώνες 10 χιλιόμετρων buffer zones δηλαδή όπου και κάποιες άλλες ζώνες όπου τα μέτρα θα πρέπει να είναι ριζικά ώστε να μην διαδοθεί προς το βορρά η ασθένεια όπου υπάρχει μεγάλη παραγωγή ε, Μεγάλε καλλιέργειε ελαιοδέντρων και να μην εξαπλωθεί αυτό προ την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό έγινε 12 Μαου, ε, υιοθετήθηκε από την Κομισιόν 12 Μαου και μετά από αυτό ζητήσαμε την Ιταλία να μα υποβάλει ένα νέο σχέδιο δράση και ειδικότερα από την περιοχή τη Πούλια. Όπω γνωρίζετε, διάφορα πράγματα λαμβάνουν χώρα στην Ιταλία ε, έγινε ένσταση κατά των μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Όπως είπατε, το Περιφερειακό Δικαστήριο έθεσε προδικαστικά ερωτήματα προς το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο στις 9 Ιουνίου ανάλυσε κατά πόσο η, το ξερίζωμα των δέντρων και στη ζώνη των 200 μέτρων τριγύρω ήταν ε, σύμφωνο με τον επιδιωκόμενο στόχο και το δικαστήριο και η Κομισιό φυσικά έμεινε ικανοποιημένη από αυτό, εκτίμησε ότι τα μέτρα ήταν αναλογικά αιτιολογημένα και μετά από αυτό ζητήσαμε από την Ιταλία να συμμορφωθεί. Η Γενική Διευθύνση Σαντέ θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα ε, με τους εκπροσώπους του ε, Ιταλικού Υπουργείου ε, Γεωργίας συναντηθήκαμε ήδη και μας εξήγησαν ότι ε, ζήτησαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο της περιοχής να συμμορφωθεί με την αποφάση του δικαστηρίου και συνεπώς να δώσει την άδεια να ξεριζωθούν, να κοπούν τα δέντρα και να λυθούν τα απαραίτητα μέτρα. Οι Ιταλικές αρχές μας εξήγησαν ότι πολλές υποθέσεις εκκρεμούσαν και ότι δεν ήξεραν πότε ακριβώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί όλο αυτό. Διότι υπήρχαν πρώτα 12 άλλες υποθέσεις, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα γίνει όλο αυτό πραγματικότητα. Εμείς φυσικά επιμείναμε να γίνει το σύντομο των δυνατόν, αλλά υπάρχουν διάφοροι κανόνες και υπάρχει και μια σειρά υποθέσεων και αυτή η υπόθεση είναι η 13η στον κατάλογο. Οι Ιταλικές Αρχές, το Υπουργείο Γεωργίας μας εξήγησε επίσης ότι πρόκειτο να, ότι μάλλον του ζητήθηκε ένα δεύτερο δείγμα για να εκτιμηθεί ότι ένα, άρθρος έχει, ένα δέντρο έχει μολυνθεί. Υπάρχουν δύο ε, δένδρα που έχουν ε, μολυνθεί στην περιοχή εξαφάνισης, ε, εξάλληψης. Μας ενημέρωσαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου πριν προβούν στην εφαρμογή των μέτρων. Κάτι που φυσικά δεν μας βρήκε σύμφωνος, διότι θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο ε, σύμφωνα με τα όσα θεωρεί η Κομισιόν. Βάσει αυτών των απαντήσεων, λοιπόν, πρέπει να σου ομολογήσω ότι απογοητευτήκαμε. Κυρίως επειδή, όπως γνωρίζετε, έχουν κατασχεθεί αυτά τα δέντρα τα οποία πρέπει να κοπούν και να εκριζωθούν και έγινε παράταση τώρα κατά 6 μήνες. Ε, από ό,τι κατάλαβαμε λοιπόν στις 13 Ιουνίου ε, έγινε παράταση κατά 6 μήνες. Κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση. Διότι τα δέντρα που έπρεπε να κοπούν δεν θα κοπούν πριν περάσουν 6 μήνες την περιοχή εξάλληψης. Ελπίζουμε στο νέο κομμάτι αυτό να γίνει γρήγορα εφόσον το Διοικητικό Δικαστήριο ε, εφαρμόσει τα μέτρα ο Επιτροπός μας θα συναντηθεί με το Υπουργείο με την κυρία Μαρτίνα από το Ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας ε, την επόμενη εβδομάδα και θα επιμείνουμε και πάλι για την υλοποίηση των κοινοτικών μέτρων το συντομότερο δυνατόν διότι όσο περισσότερο χρόνο χάνουμε τόσο περισσότερο δεν θα έχουν κοπεί δέντρα μουλισμένα και θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε το όριο της οριοθετημένης περιοχής και ένας ξέρει πού θα καταλήξει. Από πλευρά μα λοιπόν ε, ε, υλοποιούμε διάφορες ε, δικαστικές διαδικασίες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε μια πρώτη διαδικασία επί παραβάση και προετοιμάζουμε και μια νέα. Οι τοπικές τελικέ αρχές αντιμετωπίζουν ένα περίπλοκο πρόβλημα τώρα με αυτή την ποινική υπόθεση πλέον που προστίθεται. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να κάνουν ό,τι μπορούν και εμείς επίσης και η Κομισιόν δυστυχώς για αυτούς ε, θα χρειαστεί να λάβει μέτρα ε, δικαστικά επιπρόσθετα. Αυτά για την Ιταλία. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι κατάτησαν ένα σχέδιο επιτήρησης και παρακολούθησης ε, και προσέλαβαν ε, προσωπικό, αλλά αυτό το σχέδιο παρακολούθησης θα χρειαστεί τρεις-τέσσερις μήνες για να επιτηρείται σωστά η ουδέτερη περιοχή. Όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα και αργά. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ασκήσει τη μέγιστη πίεση, τη μέγιστη πίεση την Ιταλία, ώστε να δράσει. Όσον αφορά τη Γαλλία, η κατάσταση προχωρά. Υπάρχουν περισσότερες αιστείες στην Κορσική. Από όσο γνωρίζουμε είναι 253 αιστείες. Στην Προβυγγία και στην Κενιακτή έχουμε 14 αστείες. Οι γαλλικές αρχές έχουν σκοπό να εκκριζώσουν την ασθένεια. Έχουν λοιπόν ε, χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα. Έγινε ένας έλεγχος το Φεβρουάριο οι επιθεωρητές μας δηλαδή πήγαν να επιθεωρήσουν την Κωσική και την Προβυγγία και την Κιανιακτή. Η εκρίζωση ε, υλοποιείται ικανοποιητικά με τη χρήση διαφόρων ε, μεγάλων μέσων και εμείς επιμείναμε ώστε να μην υπάρξει κίνηση εκτός των μολυσμένων περιοχών γιατί δεν φαίνονταν να υπάρχουν ακριβώς στεγανά και εμείς ζητήσαμε η επιτήρηση να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γεγονός που δεν συνέβη ακριβώς, οπότε ε, στη συστάση του ελέγχου πρέπει να απαντήσει η Γαλλία. Ο Γενικός, Διευθυντή ο Γενικός Διευθυντής ε, της Γεωργίας ε, στη Γαλλία μας απάντησε είμαστε υπέρ των γαλλικών αρχών. Όλα αυτά συζητώνται κάθε μήνα στην Επιτροπή και αύριο θα το ξανασυζητήσουμε και στην ατζέντα θα συμπεριληφθούν τα διάφορα σημεία για τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία όσον αφορά τον ξυλέλο. Επίσης λάβαμε μια ειδοποίηση από τη Γερμανία στις 16 Ιουνίου για μια δάφνη που μολυνθήκε, ανακαλύφθηκε σε ένα θερμοκήπιο ιδιώτη οι γερμανικές αρχές μας ενημέρωσαν λοιπόν ότι ε, οριοθέτησαν τη ζώνη, το έχουν πάρει πολύ σοβαρά, κάνουν τις απαραίτητες έρευνες. Το σημείο συζητήθηκε αμέσως σε επίπεδο ε, φυτογειονομικών ε, διευθυντών, το συζητήσαμε, το θα το συζητήσουμε και αύριο. Για τη γερμανική περίπτωση λοιπόν ε, πρόκειται για ένα φυτό στην παρούσα φάση. Δεν μας έχουν κοινοποιηθεί άλλα μολυσμένα φυτά και ελπίζουμε να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο. Εκεί βρισκόμαστε όσον αφορά τις αιστείες στα διάφορα κράτη-μέλη. Τα μέτρα εκτέκτη ανάγκης που έχουν εφαρμοστεί από το Μάιο είναι επαρκή ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εκριζώσουν, να εξελίψουν ίσως την ασθένεια. Υπάρχει ό,τι χρειάζεται. Αλλά τώρα πρέπει να το κάνουν. Και εκεί είναι το θέμα. Τα δικά μας μέτρα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Εμείς ε, ζητάμε στην ΕΦΣΑ να ακολουθεί όλες τις νέες εξελίξεις και εμείς θα προσαρμόσουμε την απόφαση, αλλά η απόφαση ε, είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες που υπάρχουν. Έχουμε τους ελέγχους, ε, όλα τα μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως σας είπα έχουμε και δικαστικές αγωγές αυτή τη στιγμή όταν εκτιμάμε ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε. Αντιθέτως όταν κάνουν αυτό που πρέπει δικαιούνται μια χρηματοδότηση έχει οργανώσει η Κομισιόν ένα ταμείο φυτογειονομικό που μοιραζόμαστε μαζί με τους ε, ε, συναδέλφους της Ιατρικής για τα μέτρα παρακολούθησης και εκρίζωσης. Και φυσικά για να λάβει κανείς χρηματοδότηση από αυτό το ταμείο υπάρχουν συνθήκες ε, και η πρώτη συνθήκη είναι η υλοποίηση της κοινωτικής νομοθεσίας. Είναι προφανές ότι αν δεν υλοποιείται νομοθεσία τότε δεν ε, αποδεσμεύονται ε, κοινοτικά κονδύλια. Οπότε μιλάμε για ένα φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Γι' αυτό πρέπει κανείς να εφαρμόζει τα κοινοτικά μέτρα και να λαμβάνει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Από την άλλη, εκτιμάμε ότι η επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο είναι κάτι σημαντικό. Και θεωρώ ότι ο ρόλος των βουλευτών σε τοπικό επίπεδο είναι επίσης σημαντικός, ώστε να καταδεικνύει τη σπουδαιότητα ε, που, το πώς σπουδαία θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι αυτή η ασθένεια. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για όσους πρέπει να θυσιάσουν δέντρα, ε, ελιές δηλαδή, ελαιόδέντρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό είναι για το γενικό καλό, για το γενικότερο καλό της Ένωσης. Αυτό το μήνυμα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε ότι, που προσπαθούμε να διαβάσει η Κομισιόν και πιστεύω ότι και εδώ το Κοινοβούλιο έχει να παίξει κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να εξηγήσει ότι ναι μεν είναι δύσκολο για τις πληγές περιοχές αλλά ότι είναι το μόνο μέσο για να αποφύγουμε ε, σύντομα ή στο μέλλον κάποιοι άλλοι να υποχρεωθούν να πράξουν το ίδιο. Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν είναι κάτι απολύτως αναγκαίο για να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια η οποία επηρεάζει σημαντικά πιο συγκεκριμένα την παραγωγή ε, από τα ελαιόδεντρα. Εδώ αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση. Η Κομισιόν το παρακολουθεί. Μας απασχολεί όλη μέρα και εμένα και τους συναδέλφους μου. Το ίδιο και τις νομικές υπηρεσίες της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Αντρέ. Περνάμε στη συζήτηση τώρα. Η κυρία Ράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το δώρο σας. Αυτό το μπουκάλι ελαιόλαδο ε, με, το λάδι από ελιές πικουάλ. Και μάλιστα για όσους δεν το ξέρουν, σαλάτα φράουλα ή καρπούζι με τέτοιο λάδι είναι καταπληκτικό. Και είναι και χωρίς ξύλα, λέει η πρόεδρος. Ε, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα προβλήματα. Καταστροφή, ξερίζωμα, κάψιμο, μόλυνση. Ε, και μάλιστα η επιδημία ξέσπασε γιατί δεν έγιναν σωστοί έλεγχοι σε ένα λιμάνι και είχαμε μετάδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε αποφασίσει τότε να λάβουμε μέτρα για να αποφύγουμε την εμφάνιση νέων κρουσμάτων και να γίνονται πιο εντελεχείς ε, έλεγχοι στα σύνορα ε, γιατί πολύ πρόσφατα ε, τα συζητήσαμε όλα αυτά. Και μας τα υποσχέθηκε αυτά πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από ένα χρόνο επίσης επανέλαβε την ανησυχία της. Σήμερα το ίδιο. Έχουμε ένα νέο ε, κανονισμό για την φυτογεωνομική ασφάλεια για να περιορίσουμε τη μόλυνση από αρρώσχε τρίτων χωρών, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει να μειώσει τους ελέγχους στα σύνορα. Έχουμε και άλλους κινδύνους, όπως είναι ο καρκίνος των εσπεριδοειδών ή η ε, μελανή κοιλίδα. Άλλα λέει και άλλα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας υπόσχεται κάτι και ακριβώς το αντίθετο κάνει. Άλλα λέει, άλλα πράττει. Θα πρέπει, αν άλλο, να είμαστε συνεπείς και θέλουμε πραγματικά εξαντλητικούς εδελεχές τους ελέγχους στα σύνορα και να προστατευτούμε από μελλοντικέ ε, ασθένειες που θα θέσουν σε κίνδυνο την παραγωγή μας. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους ελέγχους στα σύνορα, όχι να τους μειώσουμε. Και παρόλο που μας έδωσε ως ε, αιτία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάνει λάθος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνει λάθος ε, με τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί για να υλοποιήσει το στόχο της. Χρησιμοποιεί τα αντίθετα μέσα από αυτά που χρειαζόμαστε. Και θα ήθελα να μας εξηγήσει και να μας απαντήσει την ερώτηση γιατί πιστεύετε ότι θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ασφάλεια περιορίζοντας και όχι αυξάνοντας ελέγχους ε, στα σύνορα. Η Κίνα μας ζητά 15 ε, μέρες ψυχρής ε, επεξεργασίας ε, πριν στείλουμε τα προϊόντα μας. 15 μέρες σε ψυγείο μας ζητάει η Κίνα για να στείλουμε και μάλιστα θα γίνει ο Σονούπο τα ροδάκινα και τα βερικοκάμα στην Κίνα. η Κίνα μας το ζητάει. 15 μέρες αποθήκευση σε ψυγεία. Και εμείς για να αντιμετωπίσουμε αρρώστιες όπως την, τα οματοτύπια λεοκοτρέτα, το διαβάζω όπως το βλέπω εδώ, ε, τι κάνουμε. Γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουμε παρτίδες μολυσμένες με αυτή την αρρώστια, αλλά εμείς δεν επιβάλλουμε αυτή την ανάγκη για 15 μέρες παραμονή σε ψυγεία, γιατί μόνο οι ε, ψήξη είναι αποτελεσματική αντιμετώπιση. Θα πρέπει, αν πιστεύετε ότι είναι αυτή η σωστή αντιμετώπιση, να επιβάλλουμε στις εισαγωγές αυτή τη δεκαπεθήμερη ψήξη για να αποφύγουμε περαιτέρω μόλυση. Η Κίνα απαιτεί μια τέτοια προϋπόθεση. Η Ιαπωνία το ίδιο. Εμείς γιατί μένουμε πίσω, γιατί δεν απαιτούμε αντίστοιχη προφύλαξη. Θα πρέπει να αυξήσουμε, όχι να μειώσουμε τους ελέγχους στα σύνορα. Ή λοιπόν θα αλλάξουμε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αλλιώς ξεχάστε την θεραπεία από την ξηλέλα. Και όχι μόνο δεν θα εξαλείψουμε την ξυλέλα, αλλά θα έχουμε και τον καρκίνο των εσπεριδοειδών και την μελανική λίδα και την τελευταία αρρώστια που σας είπα, λεοκοτρέτα. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρανς. Ο κύριος Σεβαστιά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ συμβολικό που μας ε, χαρίσετε ένα μπουκάλι ελαιόλαδο ακριβώς τη στιγμή που συζητούμε την ξυλέλα. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, μια ποιοτική παραγωγή. Το δώρο αφορούσε το επόμενο σημείο, την αποστολή που κάναμε στην Ανταλουσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας διαβεβαιώ πάντως ότι το ελαιόλαδο που σας χάρισα δεν έχει ξυλέλα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκπρόσωπο της ε, DG Sante, αλλά δυστυχώς δεν με καθησύχασε καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί βλέπουμε ότι οι τρεις χώρες έχουν πληγεί και σε μια ενιαία αγορά που προβλέπει ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, δεν μπορούμε, είμαστε ανίκανοι να εφαρμόσουμε μια νέα λύση και τελικά επαφιόμαστε και πάλι στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών για την εφαρμογή των μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που παρεμποδίζονται από τα δικαστικά προβλήματα που διαπιστώσαμε στην Ιταλία. Και αυτό είναι ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδυναμίας της Ευρώπης. Γιατί αν δεν είμαστε συνεπείς ε, και δεν ενισχύσουμε την απάντησή μας, δεν θα τα καταφέρουμε. Γιατί έχουμε ενιαίο πρόβλημα, ενιαία αγορά, θα πρέπει να έχουμε και ενιαία λύση. Αλλιώ το πρόβλημα θα εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Και το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι μεμονωμένο πρόβλημα των χωρών που έχουν προσβληθεί. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί και αμήλικτοι και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο ανοχής, ούτε ελευθερία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τα μέτρα που κρίνουν απαραίτητα. Πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα παντού. Και θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα από την είσοδό του. Γιατί από τη στιγμή που εισαχθεί το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο δύσκολη η καταπολέμηση του μετά. Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί είτε γιατί μερικοί αμελούν, είτε γιατί έχουμε κλιματικές αλλαγές και αύξηση της ε, θερμοκρασίας και αρρώστιες που είχαν εξαφανιστεί, που φανταζόμασταν ότι ε, δεν θα εμφανίζονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς έρχονται. Θέλουμε καλύτερη αντιμετώπιση ε, των φυτογειονομικών προβλημάτων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα πρόσχημα και μέσω ενός ε, εναλλακτικού σχεδίου θέλει να μειώσει τους ελέγχους στα σύνορα παρόλο που επίκενται και άλλες απειλές όπως ε, το black spot, ε, η μελανική λίδα ή ο καρκίνος των εσπεριδοειδών. Θα αντιμετωπίσουμε παρόμοια προβλήματα και στις καλλιέργειες αυτές, αντίστοιχα από αυτά που έχουμε τώρα με την ξυλέλα. Μία ερώτηση λοιπόν προς την Γενική Διεύθυνση Υγείας. Τι πραγματικές δυνατότητες συντονισμού έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα εξασφαλίσουμε ενιαία συντονισμένη δράση σε όλες τις περιοχές που έχουν προσβληθεί από την ξυλέλα. Επίσης, αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να σταματήσουν οι εισαγωγές από μολυσμένες περιδοδοί, γιατί ήδη έχουν διαπιστωθεί μολυσμένες σπεριδοειδή. Πού βρισκόμαστε ως προς αυτό, τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριο Τσούλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε τη Γενική Διευθύνση ΣΑΝΤ. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια εκ μέρου τη συναδέλφου Ρόζα Νταμάντο που επειδή είναι βουλευτή τη Πούλια θέλει να γίνει κάτι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ξηρέλα φαστιδιόζα και να βρεθούν βιώσιμα και αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ε, ξύρανσης, της γρήγορης ξύρανσης. Πρώτα απ' όλα, επειδή είχε εμφανιστεί σε τρία κράτη-μέλη και κοινοποιηθεί, υπογραμμίζω, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανεπίσημα σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό διότι οι εντατικές εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ, συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών ε, οδηγούν σε κυκλοφορία ε, μεγάλων ποσοτήτων βιολογικού υλικού. Οπότε μπορούμε ήδη να θεωρήσουμε ότι είναι ενδημικός οργανισμός σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στην Πούλια που έχει δηλωθεί ως μολυσμένη ε, περιοχή. Η συνάδελφος Ρόζα Ταμάτο έκανε αυτό το είδημα πριν από μήνες ε, το να αλλάξει η κατηγορία και μόνο τώρα η Κομισιόν μελετά το πέρασμα της Ξυλέλα στο παράρτημα της ε, Οδηγίας 2029 όπου ε, παρατίθεται οι οργανισμοί που υπάρχουν ε, στην κοινωτική επικράτεια. Μας αρέσει αυτή η αλλαγή πορείας, αλλά αυτό θα πρέπει να συνεπαγείται και διαφορετικά μέτρα όπως έγινε παλιότερα με την Αντρόζοφλα που είχε επιτεθεί και στην Ιταλία. Κατά την απόψή μας, η ξυλέλα δεν ε, καταπολεμάται πλέον με την εκρίζωση των δέντρων. Πρέπει να θεραπευτούν τα δέντρα από το εσωτερικό για να γίνουν πιο ανθεκτικά και αν είναι δυνατόν να σκοτωθεί το βακτήριο. Για τον λόγο αυτό, ε, μια δεύτερη σκέψη, να εστιάσουμε τις προσπάθειες στην εναλλακτική έρευνα, όπως ονομάζεται. Μέχρι στιγμής έχουμε ακολουθήσει μόνο μία οδό, την επίσημη έρευνα που διεξάγεται ε, μόνο από τον οργανισμό του Μπάρι, όπου διάφοροι εμπειρογνώμονες ε, ε, ε, ανακρίνονται αυτή τη στιγμή για την υπόθεση της ξυλέλα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Αν η Κομισιόν θέλει πραγματικά να καταπολεμήσει τη διάδοση της ξυλέλα, πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να το κάνει χωρίς τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Ε, ένα σωρό γεωργοί ζητούν αυτή, εδώ και μήνες βοήθεια γιατί βλέπουν τη δουλειά μιας ζωής να απειλείται με κρίζωση Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβει μια σαφή θέση, να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενθαρρύνει ε, εναλλακτική βιολογική έρευνα που θα βρει άλλες λύσεις ε, από την εκρίζωση των ε, φυτών. Το πρόγραμμα Horizon 2020 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς. Είναι ένα δεσμευτικό πρόγραμμα από συμμετοχής το οποίο ε, ακολουθεί τις ίδιες οδούς. Αντιθέτως, και εδώ είναι το τρίτο μου σημείο, πρέπει η Κομισιόν μέσω των οργανισμών, του οργανισμού που έκανε τη μελέτη για την ξυλέλα, να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα, να ζητήσει από την ΕΦΣΑ ε, να ενθαρρύνει τη βιολογική διαδικασία και να βρει μια εναλλακτική λύση από αυτή τη εκρίζωση των δέντρων. Ευχαριστώ κύριε Τσούλο. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, γνωρίζετε σίγουρα, εμείς ζητήσαμε την οργάνωση αυτή της ζήτησης, γιατί πραγματοποιήσαμε ημερίδες μελέτης στην Νότιο Ιταλία, στην Απουλία, πήγαμε και στην Ούμπρια, που θεωρείται η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Ελαιολάδου. Και από το πρώτο κρούσμα του Οκτωβρίου του 2013 ε, στην πουλια του βακτηρίου ξυλέλα φαστιδιώσα έχουν καταστραφεί 60.000 εκτάρια ελαιώνων. Και έχουμε πολλές οικονομικές αλλά και άλλες συνέπειες. Συναντήσαμε ερευνητέ, παραγωγούς, πολιτικούς ηθήνοντες και τους εκπροσώπους ενός γεωργικού συνεταιρισμού. Και από τις συζητήσεις προέκυψαν ε, σαφέστερα ερωτήματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 10 αλλά και η Ιταλική απόφαση έλαβαν την σοβαρή απόφαση να ξεριζώσουν τα δέντρα σε μια περίμετρο 100 μέτρων γύρω από τα άρρωστα ελαιόδεντρα ενώ οι ερευνητές λένε ότι δεν επηρεάζει ε, το βακτήριο αυτό ούτε την ελιά ούτε την περαιτέρω παραγωγή ελαιολάδου δεν επηρεάζει καθόλου την υγεία της ελιάς, ούτε αλλοιώνει ή νοθεύει την παραγωγή. Μόνο το ξύλο χτυπά. Και αν συνεχιστούν οι, ξεριζω... δέντρων, θα καταρρεύσει η οικονομία της περιοχής. Πολλό δε μάλλον που έχουμε 35.000 επιπλέον ποσόστοση ελαιολάδα από την Τινησία και μάλιστα αδασμολόγητη εισαγωγή ελαιολάδα από την Τινησία. Αν εμείς ξεριζώνουμε τα δέντρα μας και ταυτόχρονα εισάγουμε ελαιόλαδο, πιστεύετε ότι περιβαλλοντικά είναι βιώσιμη μια τέτοια λύση, για να μην σας μιλήσω για το οικονομικό. Ε, οι γεωργοί μας το επισήμαναν. Ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε το ερευνητικό κέντρο του Μπάρι. Γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί τα, τα απορίσματα της έρευνας αυτής και γιατί δεν έχει κανένας πρόσβαση στη σχετική μελέτη. Είναι απίστευτο. Φαντάζομαι οι Ιταλοί θα σας αναπτύξουν περαιτέρω αυτό το πρόβλημα που πλήττει ιδιαίτερα την Πούλια, αλλά και στη Γαλλία παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις αυτού του βακτηρίου της ξυλέλα και ε, έχουν πληγεί ελαιόδοδρα στην Κορσική και στην Προβυγγία. Ίσως ε, πιο παραδοσιακές μέθοδοι θα ήταν η λύση και όχι το ξερίζωμα των δέντρων. Σας ευχαριστώ κύριε Λόζο. Δύο μιλητές έχουμε ακόμη στον κατάλογο. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα μας είπε η συναδελφός μας για την εισαγωγή φυτών αλλά και ζώων. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά το τι εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς όπως είπε η κυρία Εράνση. Αλλιώ θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Όμω αυτά που ακούω μου φαίνονται λίγο περιπετειώδη, και ακόμα και το τελευταίο που είπε ο κύριο Ρουσό, διότι επιστημονικά είναι πολύ ξεκάθαρο τι πρέπει να γίνει. Όταν εμφανίζεται, εμφανίζεται σποραδικά κάποια ασθένεια, είτε σε φυτά είτε σε ζώα, πρέπει τα φυτά να εκριζώνονται και να καταστρέφονται και τα ζώα πρέπει να καταστρέφονται το ίδιο. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος. Γνωρίζουμε καλά τι συνέβη στην απουλία, ότι στην ουσία πρόκειται για μια διαμάχη κομμάτων, η οποία διαμάχη φάνηκε καθαρά και στην σημερινή συζήτηση. Δεν πρόκειται διόλου για επιστημονικά δεδομένα. Αυτά που ακούσαμε δεν έχουν καμία σχέση με επιστήμη. Αν θέλουμε να εμποδίσουμε την πανευρωπαϊκή διάδοση της ασθένειας αυτής και επομένως να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά η ευρωπαϊκή ελαιοκαλλιέργεια, θα πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανακόψουμε την πορεία της ασθένειας η οποία βεβαίως ανησυχεί τους ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή όπου έχει εμφανιστεί. Βεβαίως και πρέπει να απομονωθεί εκεί, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα των ε, ελαιοκαλλιεργητών, αλλά τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανακόψουμε την πορεία της ασθένειας, να την περιορίσουμε εκεί και να καταστρέψουμε τα φυτά που έχουν ε, πληγεί. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά μονάχα περιεχόμενο πολιτική συζήτηση. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για προγράμματα έρευνας που είναι απολύτως χρήσιμα και σκόπιμα, αλλά να περιμένουμε μέχρι ότου κάτι προκύψει, το μέχρι τότε η ασθένεια θα έχει χτυπήσει όλα τα λεόδοντα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μίλησαν και ευχαριστούμε και την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει η κυρία Αγγιλέρα και υπενθυμίζει σε όλους ότι το ιταλικό λάδι δεν έχει να κάνει με την ξυλέλα. Το λάδι γίνεται από ελιές ε, στις οποίες ε, δεν ε, μεταβάζεται, δεν στο λάδι ή ξυλέλα. Ευχαριστώ τον συναδελφό που το υπενθύμισε. Τρία πράγματα. Πρώτον, συμφωνά με τα όσα είπε ο κύριος ε, Ντόφμαν, και οι υπόλοιποι συναδελφοί. Το πρόβλημα είναι ότι η παγκοσμιοποίηση παγκοσμιοποιεί και τις ασθένειες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το είχαμε δει με την ασθένεια των φοινικόδεντρων και όλα αυτά. Ε, πιο πολύ έλεγχη λοιπόν στα σύνορα, διότι η στην Διώσα, όπως είπε η Κομισιόν, μπήκε αυτό το βακτήριο καραντίνας με τα ε, καλοπιστικά φυτά καφέ από την Ονδούρα και από την Κολομβία. Αναμφίβολα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα συνοριακού ελέγχου των μολυσμένων φυτών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μειώνοντα του ελέγχου, αλλά αυξάνοντά του τους ελέγχου στα σύνορα. Δεύτερον, απευθύνομαι στην Κομισιό Καταλάβετε συναδελφοί. Μιλάμε για αιωνόβια δένδρα. Ε, ήρθαν συνάδελφοι σε μια επίσκεψη στην Πούλια πριν μερικά χρόνια στο πλαίσιο τη Επιτροπή Γεωργία. Δεν είναι σαν να κόβουμε οποιοδήποτε δέντρο. Μιλάμε για δέντρα. Αιωνόβια. Ε, προφανώς Προφανώ υπάρχει και ένα κοινωνικό πολύ περίπλοκο πρόβλημα. Οπότε δείξτε κατανόηση. Έχουμε τώρα ε, κανόνε. Αλλά αγαπητοί φίλοι, ε, και το ζητώ ταπεινά από την Κομισιόν να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια ελπίδα στην περιοχή. Δεν μπορούμε να πάμε στην περιοχή του Λέτσε, στην μολυσμένη περιοχή, στην περιοχή όπου οι ευρωπαϊκοί κανόνε ε, εκ των πραγμάτων δεν εφαρμόζονται και δεν υπάρχει υποχρέωση εκρίζωση. Α προσπαθήσουμε να δώσουμε λοιπόν μια ελπίδα στου γεωργού εκεί. Τώρα η έρευνα που ενθαρρύνουμε δίνει κάποια ελπίδα για τι ανθεκτικέ ποικιλίε που δίνει τη δυνατότητα μεταφύτευσης ε, αυτών. Ε, είναι η μόνη ελπίδα που μπορούμε να δώσουμε για την ανάπτυξη της Γεωργίας. Διαφορετικά ε, καταδικάζουμε την περιοχή αυτής της Ιταλίας και τον τομέα αυτόν που είναι σημαντικός για την τοπική οικονομία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αποκριθούμε με τρόπο φυσικά αποτελεσματικό, όπως λέει η Πρόεδρος Μαρτίνα, και να τηρήσουμε τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, αλλά να εντείνει η Ευρώπη τους ελέγχους στα σύνορα να δείξει μια ελάχιστη κατανόηση όσον αφορά την εφαρμογή ενός σχεδίου που είναι πολύ ριζικό στην ουδέτερη περιοχή και ας προσπαθήσουμε να δώσουμε και μια ελπίδα για το μέλλον μέσω ε, της φύτευσης ποικιλιών που φαίνονται πιο ανθεκτικές σε αυτό το βακτήριο. Σας ευχαριστούμε κύριε Δεκάστρο. Θα ξαναδώσω το λόγο για να ολοκληρώσουμε στην εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΤΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να δώσετε κάποιες απαντήσεις γιατί είδατε πόσο έχουμε ανησυχήσει από την κατάσταση αυτή. Ελπίζω να μας δώσετε απαντήσεις και κάποιες ελπίδες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους σας για την ε, ζωηρή αυτή συζήτηση. Τι να πω, η συνοριακή έλεγχη είναι προφανές ότι η αφετηρία του προβλήματος βρίσκεται εκεί. Καμιά φορά βέβαια τα συμπτώματα δεν είναι ορατά και ούτε είναι τόσο απλό Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη ζώνη των 100 μέτρων όπου ε, αφαιρούνται τα φυτά τα οποία δεν έχουν ακόμα δείγματα της ασθένειας. Και γίνονται και εξετάσεις, τεστ πιο εξειδικευμένα που επιτρέπουν να εντοπιστεί το βακτήριο έστω και αν δεν είναι ορατά τα συμπτώματα. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2015 μετά από ψήφο των χωρών μελών απαγόρευσε την εισαγωγή φυτών καφέ. Φυτών καφέ. Που προέρχονται από Κοσταρίκα και ονδούρα. Καθαρή απαγόρευση. Επίσης για τους ε, συνοριακούς ελέγχους δεν έχουν μειωθεί. Θα πρέπει να ενισχυθούν. Είναι σημαντικό. Αυτό απορρέει και από το νέο κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα φυτά. Είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο. Άκουσα στη συζήτησή σας ότι οι εξωαγωγές μας πρέπει να υφίστανται κάποια επεξεργασία με ε, ψύχος, ε, με ψήξη δηλαδή, το ίδιο για τις εισαγωγές, μιλήσατε για τη μελανή κοιλίδα των πορτοκαλιών. Πρόκειται για ασθένειες οι οποίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο ε, κοινοτικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές και το γεγονός ότι τα ίδια αυτά κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οριοθετημένη ζώνη, δεν θα πρέπει να εξέρχονται τις οριοθετημένες ζώνες εκτός υπό πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, με αυστηρό έλεγχο. Πάντως ο κανόνας είναι ότι δεν επιτρέπεται να εξέρχονται. Εάν το συγκεκριμένο φυτόριο, για παράδειγμα, είναι μακράν ε, της ε, ζώνης που έχει πληγεί κτλ. Και ε, βεβαίως υπάρχουν επιθεωρήσεις σχετικά με τα ανθεκτικά φυτά και την έρευνα. Υπάρχουν ελαιόδεντρα που θα αποδειχθούν πιο ανθεκτικά, διότι ε, και μέσα σε ελαιόνες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ανεβρίσκονται φυτά τα οποία φαίνεται να αντέχουν, να ανθίστανται. Για το βακτήριο δεν θα αρχίσουμε να ρίχνουμε αντιβιωτικά, διότι και εσείς αν είστε άρρωστος, αν έχετε ένα βακτήριο, παίρνετε αντιβιωτικά. Διότι ε, στην περίπτωση αυτή όμως τα αντιβιωτικά ε, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο δέντρο. χρειάζονται πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης του φαινομένου και για την ώρα αυτό που υπάρχει είναι το ξερίζωμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί ορισμένα προγράμματα ερεύνης ένα πρόγραμμα του ορίζοντος 2020 που λειτουργεί, άλλο που έρχεται με διάθεση σημαντικών κονδυλίων και τα νέα προγράμματα τα οποία συζητούνται ακόμη, ανέρχονται σε 7 εκατομμύρια ευρώ για την ξυλέλα. Ελπίζουμε ότι κάτι θα προκύψει από αυτό. Και ότι πράγματι κάποια στιγμή θα είναι δυνατόν να προκύψουν ανθεκτικές ποικιλίε που θα επιτρέψουν να δοθεί και μια διαρκή λύση. Τώρα, οι ανθεκτικές ποικιλίε, όσοι, είναι, όσοι έχουν αγρονομικές γνώσεις γνωρίζουν ότι δεν είναι εύκολο αυτό, πρέπει να βρεθούν, να διασταυρωθούν, να αρχίσουν να αναπτύσσονται και ούτω καθεξής. Δεν είναι απλό δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει το γεγονός ότι πιθανώς θα είναι η λύση του μέλλοντος αυτή. Βέβαια, για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοιες ποικιλίε τουλάχιστον αναγνωρισμένες και δοκιμασμένες. Το αποτέλεσμα της ερεύνης τι να σου πω, οι ερευνητές προβαίνουν σε δημοσιεύσεις, θεωρητικά, θέλουν να δημοσιεύσουν. Ε, αυτός είναι ο στόχος των ερευνών τους. Εάν δεν δημοσιευτούν τα σχετικά αποτελέσματα των ερευνών, όπως και κάθε συνήθις δημοσίευση, ίσως διότι η δημοσίευση απορρίφθηκε από πάνελ εμπειρογνωμόνων, είτε δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα χρειαστεί λοιπόν υπομονή. Οι έρευνες διαρκούν. Οι δημοσίευση δεν είναι απλή υπόθεση. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι τα αποτελέσματα των ερευνών θα δημοσιευτούν. Γίνονται άλλωστε και προσωρινές εκθέσεις όταν οι έρευνες αυτές διαρκούν πλήωνα έτη, ε, δημοσιεύονται ενδιάμεσες εκθέσεις με αποτελέσματα. Αυτά θα γίνουν. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει για την κοινοτική έρευνα. Τώρα, οι ατομικές έρευνες, ε, αυτές δεν μπορείτε να υποχρώσετε τους ε, ερευνητές να δημοσιεύσουν εφόσον μόνο γίνουν δεκτές από κάποια επιστημονική επιθεώρηση. Το πρόβλημα για την ώρα είναι ότι είτε θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την ασθένεια και να ανακόψουμε την πορεία της ιδίως προς τον Βορρά, στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα μέτρα για την περιορισμό στην ζώνη, containment zone, δεν προβλέπουν ξερίζωμα των δέντρων. Διότι τα εγκαταλείπουν, διότι η επέκταση είναι, είναι τέτοια που αν δεν κόψουν τα πρώτα δέντρα είναι πολύ αργά. Επιμένουμε λοιπόν να κοπούν τα δέντρα γύρω στην ζώνη προστασίας όπου ακόμη δεν έχουν πληγεί στην ίδια τη ζώνη που έχει φυγεί δεν κόβονται τα δέντρα, παρά μόνο σε ορισμένες εξειδικευμένες περιπτώσεις γύρω από ένα φυτόριο, το οποίο ίσως επιτρέπεται να εξάγει ή γύρω από ορισμένες συγκεκριμένες τοποθεσίες. Όμως, ως γενικό κανόνα δεν, ως κανόνας δεν απαιτείται ε, το κόψιμο των δέντρων. Αυτές τις υποφορές μπορώ να σας δώσω. Ελπίζω ότι κάλυψα όλα όσα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι από την δική μας πλευρά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλουμε προσπάθειες και είμαστε βεβαίως διατεθειμένες να παρακολουθήσουμε τις επιστημονικές εξελίξεις, τα ενδεχόμενα άλλα μέσα που θα προκύψουν. Δεν θέλουμε να ξεριζώσουμε τα πάντα παντού. Όπως είπε ο συναδελφός σας ε, της περιφέρειας της Βόρειας Ιταλίας. Αν θέλουμε να ανακόψουμε την πορεία της ασθένειας, χρειάζεται λήψη αυστηρών μέτρων σε πολύ εξειδικευμένες ζώνες. Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος για την ώρα να αντιμετωπίσουμε το βακτήριο. Και η ΕΦΣΑ το επιβεβαίωσε. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν, διότι δεν καταστρέφουν το βακτήριο. Πρόκειται για επιβλαβή οργανισμό που έχει και σαφή οικονομική επίπτωση. Δεν είναι, δεν είναι βέβαια πρόβλημα υγείας, ανθρώπινης υγείας. Αλλά, αλλά βεβαίως εν τέλει το δέντρο αποθνίσκει. Άρα υπάρχει σοβαρή οικονομική επίπτωση. Ε, παραγωγή ελαιών αρχίζει και μειώνεται από τη στιγμή που ασθενεί το δέντρο και όταν ε, θα το κατακυριεύσει η ασθένεια θα ξεραθεί, θα πεθάνει. Άρα έχουμε κάθε συμφέρον να καταστρέψουμε το, το βακτήριο δεν έχει και προηγούμενο στην ε, Ευρωπαϊκή Φυτογειονομική Ιστορία. Ασφαλώς και πρέπει να παρακολουθείτε η εξέλιξη των επιστημονικών ερευνών, να γίνεται έλεγχος στις εισαγωγές. Όλα αυτά ωστόσο απορρέουν και από την κοινοτική νομοθεσία. Είτε λοιπόν εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε το Συμβούλιο με τους κανονισμούς βάσεως, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εκτελεστικές πράξεις. Προσπαθούμε να προβλέψουμε έναν αριθμό δράσεων. Τώρα ενδεχομένως θα υπάρχει επιτόπου κάποια αντίσταση. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ δύσκολο και ιδίω για αιωνόβια ή περαιωνόβια δέντρα που πραγματικά κλαίει η υπεραιωνοβια δεντρα που πραγματικα κλαιει η ψυχη του ανθρώπου όταν τα βλέπει να καταστρέφονται. Όμως δεν υπάρχει σωστά λύση. Τουλάχιστον στο στάδιο αυτό. Άρα πορευόμαστε με τα μέσα που διαθέτουμε. Και οι χώρες μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα σε όλα τα σύνορα για να ασκεί ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ελέγχους. Δεν είναι αξιωματούχοι τη Επιτροπή οι οποίοι τρέχουν από πίσω να δουν αν γίνονται οι συνοριακοί έλεγχοι. Προσφέρουμε ένα πλαίσιο και κίνητρα για να διεξάγονται οι έλεγχοι, του οποίου πληρώνουμε βέβαια εκ των υστέρων. Ελπίζω ότι σα καθίστηκα. Και σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Σα ευχαριστούμε κύριε Αντρέ. Φαίνεται ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους και σε παράλληλους πραγματικότητες. Είπατε ε, ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα για τα εισαγόμενα προϊόντα και οι ενόχοι στις παρεμβάσεις τους ε, είπαν το αντίθετο οι ευρωβουλευτές. Ούτε, ρωτήσε, ε, ούτε απαντήσετε συγκεκριμένη ερώτηση σε Μπαστιά για το πώς θα αλλάξει η νομοθεσία στο να επιτρεπούν εισαγωγές μολυσμένων εσπεριδοειδών με την μαύρη κοιλίδα. Εν πάση περιπτώσει, η ξυλέλα ήταν το αντικείμενο της συζήτησης, αλλά το θέμα είναι πώς θα προσαρμόζουμε τη νομοθεσία ώστε να επιτρέπουμε Εισαγωγέ περιδοειδών που είναι μολυσμένα από συγκεκριμένε ασθένειε. Εμεί ε, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, δεν θα σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση, γιατί όπω θα διαπιστώσετε και από τι παρεμβάσει, ε, μα ανησυχεί ιδιαίτερα στο θέμα. Ευχαριστώ πάντως για την ενημέρωση. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο, που ήταν και ο λόγος για τον οποίο σας μοίρασα το ελαιόλαδο. Το σημείο 12 προβλέπει την ανταλλαγή απόψεων για την αποστολή που πραγματοποιήσαμε στην Ανδαλουσία, στη γενέτειρά μου, στις 17 με 19 Μαΐου. Γι' αυτό ήθελα να σας φέρω ένα δωράκι χαρακτηριστικό από την πατρίδα μου, την Ανδαλουσία, από τη Χάεν, μια επαρχία με πολλούς ελαιώνες, όπως είναι χαρακτηριστικό και για την Νότια Ισπανία και για την Νότια Πορτογαλία αλλά και για την Νότια Ιταλία. Έχουμε πολλά ελαιόδεντρα εκεί, πολλούς ελαιώνες και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα αναμνηστικό από την ΧΑΕΝ, από τον Ελαιώνα Σεγούρα και μάλιστα από ε, ελαιόλαδο από ορεινή ε, παραγωγή. Και φυσικά είναι αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Και τώρα να σας ενημερώσω για την αποστολή που πραγματοποιήσαμε στην Ανταλουσία, Την ε, δική μου περιφέρεια που είναι μια αυτόνομη περιφέρεια της Ισπανίας ε, και από τις πιο πυκνοκατοικημένες και με το μεγαλύτερο πληθυσμό και ταυτόχρονα με μεγάλη έκταση, αντίστοιχη με αυτή της Πορτογαλίας. Έχουμε 8.300.000 κατοίκους στην Ανταλουσία το 25% επίσης της, τελικής ε, γεωργικής, της συνολικής γεωργικής ισπανικής παραγωγής. Ήταν σημαντικό να πραγματοποιήσουμε αυτή την ε, αποστολή στην Ανταλουσία. Επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος Εκέρσκι. Ε, είχαμε αρκετά πολύ μεγάλη προσωπία και Καλύψαμε σχεδόν με τις επισκέψεις μας ε, πολλές παραγωγές. Βέβαια το φάσμα των παραγωγών στην Ανταλουσία είναι ευρύτατο. Επικεντρωθήκαμε σε μερικές από αυτές για να εξοικειωθούμε με τη γεωρική πραγματικότητα της Ανταλουσίας που είναι μια περιοχή που επηρεάζει αποφασιστικά το καθάριστο χώρο προϊόν της Ισπανίας. Ξεκινήσαμε ε, με τη Σεβίλη. Εκεί πήγαμε στους οριζόνες κοντά στο, ε, στον Εθνικό Δρυμό της Δονιάνα, στο ποτάμι Γουαδαλκεβίρ. Ε, είδαμε πώς καλλιεργείται το ρύζι, γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η καλλιέργεια ρυζιού στην Ανταλουσία. Είδαμε τους οριζόνες και διαπιστώσαμε πώς συνυπάρχει η οριζοκαλλιέργεια πολύ κοντά σε έναν εθνικό δρυμό. Επίσης επισκεφτήκαμε την επαρχία της Κόρδοβας και εκεί είδαμε ένα οικοσύστημα που είναι πολύ σημαντικό στην Ανταλουσία και μπορεί να μην το γνωρίζουν όλοι. Και οι βουλευτές και η γραμματεία είδαν με τα μάτια τους ένα μοναδικό οικοσύστημα ε, που παρατηρείται στην Ανταλουσία, την Καστίγια και την Εστρεμαδούρα. Πρόκειται για το σύστημα ΔΕΕΣΑ, ένα είδος εκτεταμένου λιβαδιού, στο οποίο συνδυάζονται ε, γεωργικές, κτηνοτροφικές και δασοκομικές δραστηριότητες. Αυτή η συνύπαρξη γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοκομίας σε αυτά τα εκτεταμένα λιβάδια της ΔΕΣΑ στην Ισπανία έχει πρόβλημα ένταξης και πλαισίωσης ε, στην κοινή γεωργική πολιτική. Ακριβώς αυτού του συνδυασμού οργές κτηνοτροφίες και δασοκομείας. Γι' αυτό δύσκολα πετυχαίνουμε την αναγνώριση αυτού του συστήματος, του μοναδικού αγροδασοκομικού ε, οικοσυστήματος. Η κτηνοτροφία γίνεται ε, ελεύθερη, είναι ελευθέρας βοσκής και έχουμε κτηνοτροφία ε, προβάτων, <clears throat> βοηδών με εκτατικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτου σχεδόν ελευθέρας βοσκή στα ζώα και είναι μοναδικό αυτό το οικοσύστημα της ΔΕΣ αυτό των λιβαδιών και γι' αυτό είχε μεγάλη σημασία και συμβολικό χαρακτήρα αυτή η επίσκεψη της αντιπροσωπείας γιατί τέτοιου είδους οικοσυστήματα με εκτατική κτηνοτροφία και με συνδυασμό γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών δραστηριοτήτων είναι κρίμα να μην καλύπτεται με όλες τις τις ιδιαιτερότητες ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία και να αποκλείεται από τις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα. Είναι πραγματικά κρίμα. Και η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανταλουσίας, την οποία ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία που είχαμε και για όλη την προετοιμασία που έκανα σε συνεργασία και με την κεντρική κυβέρνηση για να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτη η αποστολή ε, μας έδωσε πολύ χρήσιμα στοιχεία. Επίσης πήγαμε σε ένα συνεταιρισμό που συγκεντρώνει όλους τους κτηνοτρόφους της επαρχίας αυτής και των γειτονικών επαρχιών της περιφέρειας. Πάνω από 3.000 κτηνοτρόφοι είναι μέτοχοι αυτής, αυτού του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού. Και μάλιστα μας είπαν κάτι που μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Μας είπαν ότι η τιμή του λίτρου γάλακτος παρά τη γαλακτοκομική κρίση δεν μειώθηκε κατάφεραν να, να παραμείνει σταθερό ε, και στα 32 λεπτά το λίτρο. Χάρη στη συσπήρωση αυτών των κτηνοτρόφων στο συνεταιρισμό. Κοβάπ είναι το όνομα του συνεταιρισμού και έχει σημειώσει πολύ πρόοδο το τελευταίο καιρό. Και μάλιστα σε μια αρχικά περιοχή με χαμηλή ανάπτυξη και με αγροτουρισμό κατάφερε να αναζωογονήσει την περιοχή και να αποκτήσει ιδιαίτερη ισχύ. Επίσης, πήγαμε και σε μια προκυπευτική ζώνη, κοντά και πάλι στον ποταμό Γοδαλκιβίρ. Εκεί είδαμε τι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για, για τα εσπεριδοειδή και τα πυρηνόκαρπα φρούτα. Και στη συνέχεια πήγαμε σε ένα κτήμα σε ένα αγρόκτημα στη Σεβίλη που είχε και ελαιόνα και εκεί κάναμε μία ανάλυση της κατάστασης ε, της ελαιοργίας. Αυτή τη στιγμή η συγκέντρωση της προσφοράς που έλαβε χώρα στην ε, Ισπανία γενικά και στην Ανταλουσία ειδικότερα έχει αποδώσει καρπούς. Ε, και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή η συγκέντρωση σε οργανώσεις ε, και σε συνεταιρισμούς έχει συμβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη και στην καλύτερη εμπορευματοποίηση των προϊόντων της ελιάς στην Ανδαλουσία. Είναι πολύ χρήσιμος ο ρόλος λοιπόν της οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα αυτό και το έργο των συνεταιρισμών πολύ σημαντικό. Επισκεφτήκαμε και ένα μνημείο, σημαντικό μνημείο της πατρίδας μου, το τζαμί της Κόρδοβα. Ε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε όλη την Ανταλουσία γιατί είναι πολύ εκτεταμένη ζώνη. Ε, και έχει πολλούς τομείς γεωργικούς. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο λιβάδι, την ΤΕΣΑ, την εκτατική κτηνοτροφία, τους ελαιώνες και την οποροκαλλιέργεια. Επίσης είδαμε και τους ε, οριζόνες γύρω από τον Εθνικό Δρυμό της Δονιάνα. Επισκεφτήκαμε ένα μικρό μέντημα της Ανταλουσίας, ε, μια περιοχή που παραλαμβάνω ότι προσωπεύει το 25% του καθάριστου εγχώριου προϊόντο της Ισπανίας. Μου υπενθυμίζει ο Φιλίππ ότι ήδη στείλαμε την επιστολή με την ενημέρωση για την αποστολή και τις δυσκολίες αυτού του οικοσυστήματος της ΔΕΣΑ για να συμπεριληφθεί στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Σας στείλαμε εμπεριστατωμένη επιστολή με υπογραφή του Πρόεδρου Σικέσκη που ήταν επικεφαλής της αποστολής μας και με τους λόγους ε, ε, για τη συμπέληψη της ΔΕΣΟ στον πρώτο πυλώνα, αλλά και την ενημέρωση από την αποστολή. Και το δώρο είναι αυτό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη ΧΑΕΝ, που έχει το αραβικό όνομα Σακούρα. Αυτά και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε τα της αποστολής τώρα. Α, ξέχασα και κάτι άλλο ασυγχώρητη. Και η Γραμματεία έχει στείλει την λεπτομεριακή ενημέρωση, την έκθεση από την αποστολή. Και ευχαριστώ θερμά τη Γραμματεία για το έργο της και ο Φιλίπ και οι παρακαθήμενοι έλαβαν μέρος στην αποστολή τους. Ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά τους που ήταν ανεκτήμητη γιατί και οι δύο αλλά και η Μάγκη που είναι η αρμόδια από τους σοσιαλδημοκράτες και η Μαλέν η βοηθός μου συμμετείχαν στη διοργάνωση και φροντίσαμε με πολλές προσπάθειες να διεξαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αποστολή. Ελπίζω να εξοικειωθήκατε με τις ιδιαιτερότητες της Γεωργίας σε ένα μικρό έστω τμήμα της Ανταλουσίας. Ο κύριος Μπόκοβιτς έχει το λόγο. Ήταν και αυτός μέλος της αποστολής. Θα μας πει από πρώτο χέρι τις εντυπώσεις του. Ευχαριστώ ε, πολύ Ήθελα καταρχάς να συγχαρώ και να ευχαριστήσω εσάς, ε, τη γραμματεία, τους ε, βοηθούς, το προσωπικό της γραμματείας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τις αρχές της Ανδαλουσίας ε, που διοργάνωσαν αυτή την εξαιρετική επίσκεψη. Είδαμε τους οριζόνες, την ε, χειροτροφία, της οργανώσεις παραγωγών, τους ελαιώνες. Είναι ένα οικοσύστημα που μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, ειδικότερα η ελεύθερη ε, κτηνοτροφία βοηδών ε, και χείρων, αλλά και ο ρόλος των, των συνεταιρισμών. Το υπογραμμίζω αυτό πόσο σημαντική είναι η οργάνωση πολλών γεωργών μαζί, γιατί έτσι αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη ε, να διασφαλίσουν την ανάπτυξή τους. Μας έκανε εντύπωση πως έχουν οργανωθεί κτηνοτρόφοι, η ε, παραγωγή γάλακτος, ε, οι συνεταιρισμοί, ε, έτσι ελέγχοντας όλη τη διαδικασία από την παραγωγή μέχρι την επεξεργασία, μέχρι το τελικό δίκτυο διανομής. Ακούσαμε και ποια είναι η τιμή, η τιμή του λίτρου γάλακτος και αντιληφθήκαμε ότι είναι καλύτερη η τιμή σε σχέση με άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτό δείχνει πόσο αναγκαία είναι η οργάνωση, η συνεργασία στη Γεωργία. Ευχαριστούμε λοιπόν για την διοργάνωση αυτού του ταξιδιού και ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε τα ίδια το Σεπτέμβριο 21-22-23 όπου θα έρθει η Επιτροπή Άγκρης στη Σλοβενία. Σίγουρα κύριε Βόκοβιτς, σίγουρα στην επόμενη μας αποστολή που θα γίνει η Σλοβενία τα αποτελέσματα θα είναι εξίσου πολύ καλά. Ο κύριος Σεμπαστιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κλάρα. Ε, θα ήθελα να σας πω ειλικρινά ότι η αποστολή ήταν εξαιρετική, η φιλοξενία άψογη και η επίσκεψη πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω με την εξοικείωση να καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτές τις λειτουργίες που είναι αναπόφευκτες και που προδίδουν την απόσταση που υπάρχει μερικές φορές μεταξύ θεωρίας και πράξης ε, στη γεωργία και εκτινοτροφία. Και αυτό ενοχλεί τους παραγωγούς, ε, η γραφειοκρατία που δεν προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό κάνουμε τις αποστολές για να μειώσουμε αυτό το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης. Πήγαμε και στη, στα λιβάδια αυτά, σε αυτό το ιδιαίτερο οικοσύστημα της ΔΕΣΑ στην ε, Ανδαλουσία. Είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί γιατί είναι μεν βοσκότοπος, είναι μεν λιβάδι, αλλά ταυτόχρονα συνδυάζει και τη δασοκομεία και την γεωργία και την κτηνοτροφία και είναι σημαντικό να καλυφθεί από τον γεωργικό κανονισμό. Και μάλιστα ο ιβυρικός Λίγκας, που είναι μοναδικό είδος στην Ευρώπη και βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, προσαρμόζεται, προχωρά, αναπτύσσεται και διαβιώνει με επιτυχία σε αυτό το οικοσύστημα, σε αυτά τα ιδιαίτερα λιβάδια της ΔΕΣΑ. Και νομίζω ότι είναι χρήσιμες αυτές οι αποστολές για να λύσουμε αυτές τις ασυναρτησίες και τα κενά που υπάρχουν μερικές φορές μεταξύ του κανονισμού και της πραγματικότητας και να καταφέρουμε να ενταχθούν και αυτά τα λιβάδια ιδέες σας στις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα γιατί είναι κρίμα να στερούνται ενισχύσεων τέτοια μοναδικά οικοσυστήματα. Πολύ χρήσιμη αποστολή και σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε κυρία Σεμπαστία. Η κυρία Μόη έχει το λόγο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την οργάνωση αυτής της αποστολής εσάς και για την υποδοχή που μας επιφυλάξαν. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο διαθέσιμοι όλοι οι άνθρωποι που συναντήσαμε και πόσο διαθέσιμοι ήταν να, να μιλήσουν μαζί μας, να μας ε, παρουσιάσουν όλη αυτή την πραγματικότητα που πήγαμε να επισκεφθούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία, διότι μετά από τόσες πολλές ε, συνεδριάσεις εδώ στην Επιτροπή Άγκρη καταφέραμε να δούμε και μια πραγματικότητα όπως έχει στην πράξη, μια καθημερινότητα όπου παρά την κρίση που χαρακτηρίζει όλη την ε, Ευρώπη στον τομέα των γαλακτοκομικών αυτή η επίσκεψη μας έδειξε πόσες δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν ένα υπόδειγμα όπου υπάρχει προστασία και παρακολούθηση σε όλα τα βήματα της αλυσίδας της παραγωγής από τους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές μέχρι το τελικό προϊόν. Και όπως είδαμε είναι μία από τις ε, περιοχές, ε, τις λίγες, ε, όπου δεν μειώθηκε η τιμή του γάλακτος. Υπήρχε προστασία δηλαδή για τους παραγωγούς κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη με την κρίση που ε, αντιμετωπίζουμε. Ήταν λοιπόν ένα άριστο παράδειγμα του πώς μπορεί να διοργανωθεί καλύτερα ο όλος τομέας, ολόκληρη η παραγωγή. Ήθελα επίσης να επισημάνω κάτι ενδιαφέρον, το οποίο αντελήφθηκα συζημινομιλώντας με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Είναι η πτυχή της συνεργασίας η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, από τον παραγωγό κτηνοτρόφο μέχρι τα ερευνητικά κέντρα, με ειδικευμένο προσωπικό που τους βοηθούν να συλλέξουν και κονδύλια από την Ευρώπη και όλη αυτή σε συνεργασία με τις ιδιωτικές εταιρείε. Είδαμε δηλαδή μια εξαιρετική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, άψογη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που όταν χρησιμοποιούνταν για την έρευνα, ε, τα αποτελέσματα ε, εφαρμόζονταν μετά, αξιοποιούνταν στην ε, περιοχή, ώστε να παρέχουν μια αξιοπρεπή ζωή ακόμη και στους μικρότερους συμμετέχοντες ή παραγωγούς, παρά την κρίση και παρά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί στην Ευρώπη συχνά αποκομίζουν όλο το κέρδος η μεγάλη παραγωγή εις βάρος των μικρών παραγωγών, ενώ σε αυτή την περίπτωση είδαμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ε, πράγματι θα έπρεπε να λειτουργούν ε, οι διαδικασίες παραγωγής στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ και τη συναδέλφη την κυρία Αγγελίερα. Σας ευχαριστούμε κυρία Μόη. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Αυτός ήταν ο στόχος, ε, να σας δώσουμε μια γεύση για την πραγματικότητα της Ανταλουσίας. Και με χαροποιούν τα σχόλιά σας γιατί μου δείχνουν ότι πραγματικά καταφέραμε το στόχο μας. Επιτύχαμε το σκοπό μας και ευχαριστώ τη Φιλίπ, τη Μαλέν, τη Μάγκη, όλους ε, όσοι έλαβαν μέρος στην αποστολή και όσους βοήθησαν να, ε, να στεφθεί με επιτυχία. Η επόμενη μας αποστολή θα γίνει το Σεπτέμβριο στη Σλοβενία, στην πατρίδα σας κύριε Μπόγκοβιτς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, και είμαι βέβαιη ότι και η αποστολή εκείνη θα είναι αίσια. Περνάμε τώρα στο σημείο 13, την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Στην χθεσινή συνεδρίαση, χθε το πρωί, οι συντονιστές κατέληξαν σε συστάσεις που σας τις στείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τις έχετε λάβει και σε έντυπη μορφή. Αν θέλετε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, παρακαλώ μπορούμε να εγκρίνουμε τη στάση των συντονιστών. Έτσι φαίνεται, πολύ ωραία. Οπότε, αν δεν υπάρχουν διάφορα, να σας ενημερώσω για τις επόμενες μας συνεδριάσεις που θα γίνουν 19 Ιουλίου. Τέλειο δώρο κάνουμε στους εαυτούς μας. 19 Ιουλίου το πρωί έκτακτη συνάντηση με τον Επίτροπο Χόγκαν. 8.30 με 10.30 το πρωί. Ανοιχτή συνεδρίαση των συντονιστών. Και αυτοί που λένε ότι η Επιτροπή Γεωργίας ε, είναι νοθροί είτε μπέλα, πρέπει να κοιτάξουν, γιατί είμαστε η μόνη επιτροπή που έχει συναντήσει την επόμενη εβδομάδα. Και μετά τις θερινές διακοπές ε, θα ξανασυναντηθούμε στις 30 Αυγούστου 9 με 12.30 το πρωί. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές. Θα είμαι φυσικά και στην έκτακτη συνεδρία τη επόμενη εβδομάδα, αλλά και θα προεδρεύσει ο πρόεδρο. Καλό καλοκαίρι, καλέ διακοπέ, καλή ξεκούραση και να επιστρέψουμε ακμαίοι και θριαμβευτικοί το Σεπτέμβριο. Γεια σας.